Ραμπέλα, ολοκληρώνω τη συζήτηση εδώ. Η ψηφοφορία θα γίνει την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, όχι αύριο. Η επόμενη συνεδρία είναι αύριο.